Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε μια σειρά από ψηφοφορίες. Να σας δώσω λίγο χρόνο για να βάλετε την ε, κάρτα σας ε, στη συσκευή για τυχόν ηλεκτρονική επαλήθευση. Το πρώτο θέμα είναι η διαθεσμική συμφωνία σε συνεργασία ε, για θέματα προπολογισμού. Μπορούμε να περάσουμε στην τροπολογία 1, υπέρ, κατά, δεν είδα τίποτα, δεν έχετε όρεξη να σηκώσετε τα χεράκια σας σήμερα. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία.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 41 κάρτε, 39 ψηφίσατε, πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται 29, 6, 4 εποχέ. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω έχει διαγραφεί η 6, έχει αποσυρθεί η 6, συμβαστική τροπολογία 3 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1, τροπολογία 10, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορίας, 40 υπέρ, 1 κατά, 2 αποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, εγκρίθηκε η έκθεσή της. Να περάσουμε τώρα. Μισό λεπτάκι, διότι πρέπει να έρθει στο γραφείο της Προεδρίας ο υπάλληλο που παρακολουθεί το θέμα. Για την ψηφοφορία μας, ε, το θέμα είναι πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία σε ανάπτυξη πολιτικο-στρατιωτικών ικανοτήτων. Η συγγήτρια κυρία Έλερ. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 που είναι συμβατή με τη συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21, υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 21, όχι 11. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά δεν είμαι βέβαιος, να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. 44 κάρτε, 44 κάρτες, 43 ψηφίσαντες, Πέρας της ψηφοφορίας, 32 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. 46 και 46 46 ψηφίσαντες πέρας της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται. Ναι. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. al 33. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 38 δεν ψηφίζεται γιατί είναι απλώς ε, γλωσσική διαφορά. Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, να κάνουμε όμως ε, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 59. 47. 47 ψηφίσατε πέρα τη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 60 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, Ζητώ συγγνώμη, όπως πολύ σωστά μου επισημαίνουν, έκανα λάθος εγώ, πρέπει να ψηφίσουμε την 62 γιατί απορρίφθηκε η 61. Ψηφίζουμε λοιπόν την 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 77 αποσύρεται, η 81 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, Αποχές εκρίνεται 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να περάσουμε τώρα στην 78. Λοιπόν, απορρίψαμε το δεύτερο τμήμα τη 81, επομένω πρέπει να ψηφίσουμε την 82. Ψηφίζουμε λοιπόν την 82. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78. Υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 79. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επειδή απορρίφθηκε η 89, θα ψηφίσουμε την 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές είχε ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία για την 107. Έχει γίνει αποδεκτή. Ωραία. Θέλει κάποιος από τους πρασίνους να λάβει το λόγο ή θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. need to have the floor. Δεν χρειάζεται να πάρω το λόγο, απλά ήθελα να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, δεν έχουμε ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε κανονικά. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 112 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε την 113 γιατί είναι ίδια. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108. Συμβιβαστική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 4 έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από ε, πλευράς ε, του ECR. Ψηφίζουμε λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία 4. Απέρτα la votazione. 49 schede, 49 votanti. 49 ψηφίσαντες, πέρας της ψηφοφορίας, 38 κατά, 11 υπέρ, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 124 υπάρχει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από πλευρά των πρασίνων. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 47 ψηφίσαντε, εγκρίνεται 34 υπέρ, 10 κατά, 3 απόχέ. το δεύτερο τμήμα αποσύρεται, συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ. Κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10, υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 134, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135, υπέρ κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το 135, η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασες ψηφοφορίας, 47 ψηφίσαντες, 34 κατά, 14 περ 0 αποχές απορρίπτεται. 136 περ Κατά, αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, άρχεται η ψηφοφορία γιατί είναι 142. «48 ψηφίσαντες πέρα της ψηφοφορίας» 27 υπέρ, 21 κατά εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική επαλήθευση για την 150. 50 σκέδι, 50 ψηφίσαντες. Απορρίπτεται.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 50 votanti. πέρα votazione. 50 39 υπέρ, 2 κατά, 9 αποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, εγκρίνεται. Επόμενο. Ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χημικό, βιολογικό, ραδιολογικό και πυρηνικό τομέα. Συντάκτρια η κυρία Λούσινγκ. Τροπολογία 26. Υπέρ.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 Ο τίτλος που σας είπα είναι σωστός, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, μισό λεπτό γιατί... Va bene, va bene. Allora, possiamo procedere. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Ε, γνωμοδότηση της κυρίας Λέζινγκ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 4, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, Παρακαλώ, κύριε Νταβί. Στον κατάλογο ψηφοφορίε προβλέπετε ότι εφόσον εγκρίνουμε την τροπολογία 1, η 3 καταπίπτει. Γιατί την ψηφίσαμε λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Eh, Σωστά, έχετε δίκιο. Το, η τρία δεν έπρεπε να ψηφιστεί γιατί είχαμε εγκρίνει την 1. Εγκρίναμε την 4. Πηγαίνουμε λοιπόν στην τροπολογία 5, υπέρ. Τροπολογία 5, υπέρ. Κατά, αποχές, αποχές, εγκρίνεται. 6, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Λοιπόν, πάμε στην τροπολογία 13 γιατί εγκρίναμε την 7, οπότε οι επόμενες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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, υπέρ,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 Από τη 15 πάμε στην 22. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται 23. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται και 25. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. 52 51 votanti. Chiusa la 51 ψηφίσαντες πέρας ψηφοφορίας, 30 υπέρ, 18 κατά, 3 αποχές εγκρίνεται. 28 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Αν δεν σηκώνετε όμως τα χέρια σας, ε, δεν μπορώ να δω το αποτέλεσμα. Πρώτο τμήμα της 28, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πρώτο τμήμα. 52 ψηφίσαντες, 33 κατά 19 υπέρ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά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 32 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση από το ΕΛΚ το αίτημα για την 33 52 κάρτες 51 ψηφίσαντες πέρασε της ψηφοφορίας 32 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Μισό λεπτό, ο κύριος δεν θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίσαμε την τροπολογία 35. Sì, e 30 33. Από την 30 περνάμε στην 33. Πέρασε η 30, επομένω οι υπόλοιπε ε, καταπίπτουν. Αυτό έχω εγώ εδώ στο κατάλογο. 38 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Συγγνώμη, 43 αποσύρθηκε. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 49 υπέρ, 2 κατά, συγχαρητήρια στη συντάκτρια. Να ψηφίσουμε τώρα τη γνωμοδότηση του κυρίου Πεγιών, χορήγηση εγγύηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύησει για σχέδια εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. aspettarlo Bene. Ε, Possiamo allora procedere. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 27 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Έχετε κάτι να πείτε. Η 66 αποσύρθηκε, η 67 ψηφίζεται. Άρα δεν έχετε τίποτα να πείτε. 67 απορρίφθηκε, συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Με την προφορική τροπολογία αριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική απολύθευση για την 74. 50 σκέδες 47 50 κάρτες, 47 ψηφίσατε, 25 κατά, 20 υπέρ, 2 αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απο, εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με την ε, προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 80 με την προφορική τροπολογία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Υπάρχει έτοιμα για ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 80. Άρχεται η ψηφοφορία. 50 schede, 49 50 votanti, chiusa la votazione. 50 ψηφίσαντες, πέρας ψηφοφορίας, 35 κατά, 15 υπέρ, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 με προφορική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 με την προφορική τροπολογία 8 υπέρ. Καταπίπτει, πάμε στη 36 υπέρ. Υπέρ τη 36. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 με την προφορική τροπολογία περιθμών 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 με την ε, προφορική τροπολογία 10. Να βάλουμε λίγο το 39, διότι οι πράσινοι ζητούν ηλεκτρονική επαλήθευση για την 91. Άρχεται η ψηφοφορία. σχέδια, 49 votanti. Chiuda chi. 50 va bene. 30. 50 33 κατά, 17 υπέρ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39 με την προφορική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 και 97 που ψηφίζονται από κοινού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 98 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 πρέπει να ψηφίσουμε τη 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 2. Άρχεται η ψηφοφορία. 50 schede, 49 votanti. 50 49 ε, ψηφίσαντες, 36 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται με αθρώα πλειοψηφία, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σας. 41 υπέρ, κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά. απόχέ. εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά. Αποχές, Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 αποσύρεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αποσύρεται 47, 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά,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 Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 με την προφορική τροπολογία υπαριθμών 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος να ελέγξουμε την 64. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 64. 50 ψηφίσαντες. Πέρασε ψηφοφορίας. 42 κατά 8 υπέρ. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. 50 schede, 48, 46 48 ψηφίσατε, 46 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Ε, συγχαρητήρια στο συντάκτη τη γνωμοδότησης. Πρωτόκολλο στη Συμφωνία Εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Μολδαβίας. Μόνο την ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να κάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, έκθεση Watson. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. 49 υπέρ, κανείς κατά. Τεράστια πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Βότσον. Συγκρότηση μηχανισμού ταχεία αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάκτρια τη γνωμοδότηση κυρία Βέμπερ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 9. Α. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται, 12 υπέρ, κατά, Δεν είμαι βέβαιος. Για να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. 48 σχέδι, 47 votanti. 48 ψηφίσαντες πέρασε ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 16 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ. Α, συγγνώμη. Εγκρίναμε την 16, επομένως καταπίπτει 17. 18 υπέρ. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 18. «49 schede, 47 votanti. Chiusa. Πέραση ψηφοφορία, 47 ψηφίσαντες, 34 κατά, 10 υπέρ. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση για την 21. Πολύ καλά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 21. Πέραση ψηφοφορία 22 κατά 27 υπέρ εγκρίνεται. 22 με την προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. 39 υπέρ, 8 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση συγχαρητήρια στο συντάκτη. Στη συντάκτρια μάλλον. Ένα μικρό διάλειμμα, πέντε λεπτά, για να συνεχίσουμε κατόπιν με την μερίσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη, η οποία προβλέπει την έκθεση μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Η συγητής είναι ο κύριος Αρλάκη. Ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει την ε, παρέμβασή του Τίνουμε δίκονους. Παρακαλώ κύριε Αρλάκη. Ευχαριστώ. Πρόκειται για τη συνάντηση πριν, τελευταία συνάντηση πριν από την ψηφοφορία και εντωμεταξύ έχουν κατατεθεί συμβιβαστικές τροπολογίες στην οριστική μορφή τους και υπάρχει γενική συμφωνία, ομοφωνία για ε, τις 22 συμβιβαστικές τροπολογίε. α, συγγνώμη, 26 διορθώνει ο ομιλητής, συμβιβαστικές τροπολογίες που καλύπτουν πολλά άρθρα. Θα ήθελα λοιπόν απλά στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για κάποιες εξ αυτών. Και για να εξηγήσω δηλαδή γιατί στον κατάλογο ψηφοφορίας έχω βάλει αρνητικό πρόσημο σε κάποιες περιπτώσεις γιατί υπάρχουν πολλές επικαλύψεις και υπάρχει και ένα πρόβλημα ως προς το ύφος της ε, έκθεσης. Εγώ θέλω να είναι ευανάγνωστη για όλους η έκθεση. Αποφεύγω λοιπόν κατά το δυνατόν ειδικέ εκφράσεις ή εκφράσεις που παραφορτώνουν την έκθεση. εξι 7 τροπολογίες ε, θεωρώ ότι είναι κάπως φλίαρες και επαναλαμβάνουν ε, αρχές που έχουν αναφερθεί και σε άλλα σημεία της έκθεσης. Γι' αυτό και τις έχω απορρίψει. Αλλά θα έρθω σε επαφή με τους ε, συναδέλφους που έχουν καταθέσει τις τροπολογίες και θα τους ζητήσω να τις αποσύρουν. Γιατί έχουν καλυφθεί αυτά που λένε, δηλαδή έχει κάποιον άλλο λόγο. Να πω τώρα να κάνω μια τεχνική σημείωση. Υπάρχει ένα σφάλμα μία από τις συμβαστικές τροπολογίες, στην 19 για την ακρίβεια, ως προς τον αριθμό των Αφγανών που ασχολούνται με και ζουν από τη δεδεμπόρη του όποιου. Μιλάμε για 1,6 εκατομμύρια Αφγανούς, όπως αναφέρεται και κάπου αλλού στην έκθεση. δεν είναι ο σωστό αριθμός 1,4 εκατομμύρια, είναι 1,6 εκατομμύρια για να υπάρχει κάποια συνοχή στην έκθεση. Να το αλλάξουμε λοιπόν αν θέλετε και αν συμφωνείτε. Πρωτού υποβάλλουμε και το τελικό κείμενο των συμβαστικών τροπολογιών. Η τροπολογία 306. στην, ε, στο σημείο 4. Θέλουμε να αλλάξουμε το police training σε police και security training. Και rule of law. Εγώ να προτείνω να αναφέρεται και η αστυνομία και το κράτος δικαίου. Γιατί έτσι θα καλύπτονται και οι δυνάμεις ασφαλείας, αν συμφωνεί και ο συνάδελφος που κατέθεσε την τροπολογία. Στην τροπολογία 370, 371, 372 Κασουλίτης, Γιαννάκου, Φανόρνταν, στην παράγραφο 62. Να προτείνω σε όλους τους συναδέλφους να αποδεχτούμε το πρώτο κείμενο, το αρχικό κείμενο και να αλλάξουμε το, τους συμμάχους ΝΑΤΟ σε Αφγανούς συμμάχους. Γιατί δεν είχα διευκρινίσει στην αρχή ότι ε, αναφερόμουν στους συμμάχους α, τους Αφγανούς. Άρα, να διορθώσουμε, αν θέλετε, στο αρχικό κείμενο την διατύπωση. Να αλλάξει το NATO Allies και να γίνει Afghan Allies και στην ε, τροπολογία 60, Νόιζερ και άλλοι, μία άλλη τεχνική αλλαγή για τις αγορές οποίου να πούμε αγορές ηρωίνης. Γιατί εδώ πέρα στην Ευρώπη δεν έχουμε αγορές οποίου έχουμε αγορές ηρωίνης ουσιαστικά. Αυτά λοιπόν ήθελα να διευκρινίσω. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο και να απαντήσει, να συζητήσουμε κάτι, και φυσικά, αν, θέλουμε, αν θέλετε να πάρετε το λόγο για κάποιο άλλο θέμα, εδώ είμαι. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά επειδή εσείς μου το δίνετε μόνο σας, δέχομαι και θα, θα μιλήσω. Θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε ότι ο κύριος Κασουλίδης, ο οποίος είναι ο σκιώδης εισηγητής από πλευρός της ομάδας μας, μου ζήτησε, επειδή αποσιάζει στην Κίνα, να κάνω κάποια σχόλια για την έκθεση του κυρίου Αρλάκη μετά από την ε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε. Στην Επιτροπή μας. Καταρχήν, μου ζήτησε ο κύριος Κασουλίδης να διαβιβάσω τις ευχαριστίες του προς τον κύριο Αρλάκη για το συνεργάσιμο πνεύμα και την καλοσύνη του να λάβει υπόψη μερικές από τις τροπολογίες. Όπως ξέρετε κύριε Αλάκη, το θεμελιώδη στοιχείο για την πολιτική μας ομάδα είναι να διαμορφωθεί μια ισορροπημένη έκθεση που να λαμβάνει υπόψη τη νέα στρατηγική. Και από αυτή την άποψη Αντιλαμβανόμαστε τα σφάλματα που διαπράχθηκαν στο παρελθόν και επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για μια αξιολόγηση των συνεπειών αυτής της νέας στρατηγικής κατά των, της ανταρσίας, κατά των εξεγέρσεων. Και γι' αυτό επιμένω στην ανάγκη να διασφαλίσουμε την ε, ισορροπία της έκθεσης. Ο κ. Κασουλίδης έθεσε και ορισμένα ακόμη σημεία Καταρχήν, ενώ θα πρέπει φυσικά να τηρήσουμε αυτήν την ανάγκη της ισορροπίας, καλό θα ήταν οι συμβαστικές τροπολογίες να συνδυάζουν τα λάθη του παρελθόντος με τα διδάγματα που αντλούμε από τα λάθη αυτά και να θέσουμε την έμφαση στην ανάγκη μιας πολιτικής διαδικασίας για να βρούμε λύση στα προβλήματα και την κατάσταση του Αφγανιστάν. Μια πολιτική λύση που δεν θα περιορίζεται στο διάλογο με ορισμένες φατρίες των Ταλιμπάν, αλλά ε, θα εξαρτηθεί και από την ε, στρατιωτική αποδυνάμωση των Ταλιμπάν. Κάποιοι βουλευτές της ομάδας μου θα ζητήσουν κάποια χαλάρωση της διατύπωσης για να μην υποσκάπτουμε την ίδια μας τη θέση και επίσης ε, θα προσπαθήσουμε η παγκόσμια βοήθεια που ούτως ή άλλως είναι γενναιόδορη να αξιοποιηθεί καλύτερα και να είναι πιο αποτελεσματική. Ο κ. Κασουλίδης μου είπε ότι οι δωρητές ε, και οι χορηγοί παγκοσμίω θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο δεδομένη της κατάστασης του Αφγανιστάν. Σας ευχαριστεί ο κύριος Κασουλίδης που υπογραμμίζεται τη σημασία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της καλλιέργειας του οποίου. Ξέρετε πόσο συμβάλλει η καλλιέργεια της Μύκονος Υπνοφόρου στην, και των ναρκωτικών γενικώ ε, στην ε, αύξηση του ΑΕΠ. Και φυσικά θέλουμε να προχωρήσουμε και να νικήσουμε στρατιωτικά τους Ταλιμπάν, αλλά θα πρέπει να προβάλλουμε αυτό το συσχετισμό μεταξύ του πλούτου που παράγουν τα ναρκωτικά και της ε, σημασίας που θα πρέπει να έχει η στρατηγική μας στο Αφγανιστάν. Ο κύριος Κασουλίδης Προσωπικά είναι κατά της χρήσης ε, παρασιτοκτόνων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Παρόλο που μερικοί καλλιεργητές είναι αντιδραστικοί και αρνούνται να περάσουν σε εναλλακτικές καλλιέργειες, παρόλα αυτά είναι κατά της χρήσης των παρασιτοκτόνων. Επίσης, ε, αντιλαμβάνεται ο κύριος Κασουλίδης, παρόλο που γνωρίζει τον περιορισμό που έχουμε στον αριθμό των σελίδων, πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στην κατάρτιση και την εξάσκηση των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά να δώσουμε έμφαση και στο θέμα του στρατού. Οι δυνάμεις ασφαλείας και του στρατού αλλά και της αστυνομίας θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας μέχρι το 2014. Για όλα αυτά λοιπόν κύριε Αρλάκη, θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Κασουλίδης συμφωνεί καταρχήν με τις 26 συμβαστικές τροπολογίες, παρόλο που όπως σας είπα για την τροπολογία 14 ε, θα καταψηφίσει μία παράγραφο. Αυτό που μας ανησυχεί πάντως κύριε Αρλάκη είναι το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται δεσμευθήκατε να δεχτείτε και μεμονωμένες τροπολογίες της πολιτικής μας ομάδας, αλλά από ό,τι φαίνεται από τον προκατατικό κατάλογο ψηφοφορίας, βλέπουμε αρνητικό πρόσημο σε αυτές τις τροπολογίες, παρά τη δέσμευσή σας να τις δεχτείτε. Αυτά ήταν τα σχόλια εκ μέρους του σκιώδου συγητού της ομάδας μου, του κ. Κασουλίδη. Βέβαια, έχουμε χρόνο, γιατί αν δεν κάνω λάθος θα ψηφίσουμε ή στις 8 ή στις 9 του μηνός. Επαναλαμβάνω, σας ευχαριστούμε για το διαλεκτικό σας πνεύμα και για την ε, προθυμία σας για διάλογο. Η έκθεση αυτή είναι πραγματικά κρίσιμη για μια χώρα στην οποία εκτιλήσεται πολύ σημαντικός αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Και είναι σκόπιμο να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη υποστήριξη και τη Επιτροπή μας και τη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε λοιπόν μια ισορροπημένη έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα λεπτά και ευαίσθητα σημεία και φυσικά θα πρέπει να υποδείξουμε τα λάθη και να ασκήσουμε κριτική, αλλά να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη προόδου και όχι εγκλωβισμού στα αρνητικά σημεία. Γιατί άλλο είναι η επικοδομητική κριτική και άλλο είναι να ε, υπονομεύουμε τη θέση μας, ιδιαίτερα με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοι του στο Αφγανιστάν. Αυτά λοιπόν ήταν κύριε Αλάκη τα σχόλια του κύριου Κασουλίδη και πάλι θερμά ευχαριστώ για το διαλεκτικό σας πνεύμα και την προθυμία σας για διάλογο και ευελπιστώ ότι μέχρι την ψηφοφορία θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την έκθεση που είναι πολύ σημαντική, που επαναλαμβάνω καλό θα ήταν να τύχει τη ευρύτερη δυνατή υποστήριξη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ο κύριο Στάλλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται καν να επαναλάβω το μεγάλο μου θαυμασμό και την εκτίμηση που τρέφω προς το έργο του κυρίου Αρλάκη και των σχεδόν εισηγητών. Πραγματικά είναι πολύ καλή έκθεση και πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι καλή γιατί πραγματικά κάνει μια γενική επισκόπηση της κατάστασης του Αφγανιστάν αλλά υπάρχουν και κάποιες παραλήψεις ό,τι αφορά την ενάργεια του κεντρικού μηνύματος της έκθεσης, που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε την διεξαγωγή μιας πολιτικής διαδικασίας που θα επιτρέψει το συντομότερο δυνατό, έστω και σε λίγους μήνες, μακάρι και σε λίγους μήνες, μπορεί και σε κάποια χρόνια, να επιτρέψει λοιπόν την απόσυρση των συμμαχικών δυνάμεων. Οι ψηφοφόροι μας και το κοινό υποστηρίζει ένθερμα αυτή τη στρατηγική. Ο κόσμος, ο λαός θέλει να οργανώσουμε πολιτικά τη δυνατότητα αποχώρησης των συμμαχικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Όχι από κάθε χώρα ξεχωριστά και μονομερείς αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβούλων. Αλλά το ευρωπαϊκό κοινό περιμένει μια στρατηγική συνολική, στρατηγική της συμμαχίας. Στην συμβαστική τροπολογία 13, ο κύριος Αρλάκη αναφέρει ότι η τροπολογία μου 273 καλύπτεται από προηγούμενη συμβαστική τροπολογία. Ίσως ε, δεν κατάλαβα καλά εγώ ή την έχασα κάπου την τροπολογία μου, αλλά εγώ πιστεύω ότι η τροπολογία 25 είναι πιο κοντά σε αυτό το μήνυμα προσπάθησα να μεταβιβάσω με την τροπολογία μου. Ότι δηλαδή θέλουμε στο μέλλον αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων. Δεν βλέπω σε καμία άλλη συμβαστική τροπολογία αυτό το στοιχείο. Η τροπολογία μου 273 απευθύνει έκκληση για μια διευρυμένη πολιτική διαδικασία στο Αφγανιστάν που θα περιλαμβάνει όλες τις ε, πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις του Αφγανιστάν και που θα επιτρέψει την απόσυρση των συμμαχικών δυνάμεων. Αν διαβάσουμε καλόπιστα την ε, συμβαστική τροπολογία 25, εμπεριέχει κάπως αυτό το μήνυμα. Γιατί λέει και οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμη ε, δείξει την πρόθεσή τους να αποσυρθούν, ενώ η, απο, η απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων πρέπει να έχει ένα σταδιακό και συντονισμένο χαρακτήρα και το καθεξής. Ίσως το μήνυμα αυτό θα πρέπει να καταστεί πιο σαφές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ από την ομάδα μου, ως και ο θα είμαι σύντομο. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Αρλάκη, ο οποίος ε, κατάφερε να βρει ε, ευρείε ε, συμβαστικέ λύσεις, τις οποίες στηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες και είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει με την συνένεση αυτή να δηλώσουμε ότι ενθαρρύνουμε την πολιτική εξέλιξη στο Αφγανιστάν. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη των ασφαλώς και τις νέες στρατηγικές που έχουν ε, καταρτιστεί στο Αφγανιστάν. Ίσως να υπάρχουν και κάποιες προσθήκες που θα πρέπει να γίνουν, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Τάλερ, αλλά νομίζω ότι η τροπολογία συμβαστική 25 ξεκαθαρίζει ποιο είναι το επόμενο βήμα για μας και ότι θα πρέπει μέχρι το 2014 να έχει ολοκληρωθεί ή θα πρέπει να έχει επισπευστεί η στρατηγική εχει επισπευθει η Αυτά που είπε ο συνάδελφος Αρλάκη για την ε, αστυνομία και το κράτος δικαίου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι το κράτος ε, δικαίου έχει την ίδια θέση όπως και η εκπαίδευση των αστυνομικών και σε ό,τι αφορά την διευκρίνηση ότι πρόκειται για αγορές ε, ηρωίνης και όχι οποίου, είναι σωστό και αυτό. Χαίρομαι που υπάρχουν ε, αυτοί οι συμβιβασμοί, τις οποίες υποστηρίζουν και οι ομάδες και έτσι πολιτικά νομίζω μπορούμε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Merci, Président. Κυρία ευχαριστώ. Φυσικά όταν λαμβάνει καλή στο λόγο μετά από συναδέλφους προλαλήσαντες δεν μπορεί παρά να επαναλάβει ορισμένα πράγματα αλλά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Αρλάκη για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε και για το ότι συμπεριέλαβε και αρκετές τροπολογίες δικές μου στις συμβαστικές του προτάσεις. Βέβαια, δεν συνέβη με όλες τις τροπολογίες. Θα ήθελα παρόλα αυτά να επιμείνω και να σας εξηγήσω γιατί είναι χρήσιμε οι τροπολογίες μου. Για παράδειγμα, η τροπολογία 14. Είχα ζητήσει από τον εισηγητή να προσθέσουμε μνήα του συντάγματος του 2004. Συγγνώμη, είναι η τροπολογία μου 33, όχι 14. Ή μάλλον η τροπολογία 14 για το κεφάλαιο 33. Να προσθέσουμε το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μνήμα του συντάγματος το 2004. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αναφορά του συντάγματο του 2004, γιατί όπω είπε και πριν από λίγο ο κύριο Αλαφράγκα, είναι ένα τρόπο ε, αμέσω για να επιμείνουμε και στα θετικά σημεία. Και αυτό είναι ένα θετικό σημείο. Γιατί φοβόμαστε κάποια παλινδρόμηση. Χρήσιμο λοιπόν είναι να αναφέρουμε την έκθεσή μας το Σύνταγμα το 2004. Και κάποια άλλα σημεία. Στην τροπολογία 11 για παράδειγμα. Εκεί δεν επιμείνατε στις προδιαγραφές διαφάνειας και στα κριτήρια χρήσης ό,τι αφορά την αλυσίδα ανεφοδιασμού. Καλή ε, τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο μέτρο που είναι υπεύθυνε για την, ε, αλυσίδα τους, για την δική τους αλυσίδα ανεφοδιασμού. Να αναφερθούν λοιπόν και τα πρότυπα διαφάνειας και τα κριτήρια χρήσης. Επιμένω κύριε Αρλάκη. Αυτά ήταν τα δύο σημεία. Παρ' όλα αυτά μας ε, χαροποιεί το ότι συμπεριλάβατε πολλές τροπολογίες και χαίρομαι που λάβατε υπόψη ειδικά τις τροπολογίες για την ένταξη στην κοινωνία των γυναικών του Αφγανιστάν. Η κυρία Γκόμες. Would like to thank uh, uh, Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Αρλάκη και τους σκιώτες εισηγητές για τον τεράστιο όγκο δουλειά που κάνουν. Και έτσι συμπεριλαμβάνονται πιο πολλές τροπολογίες και υπάρχει πραγματικά συνοχή στο κείμενο. Πολύ καλή η δουλειά τους. Και προφανώς αυτό χάρη είναι στο ανοιχτό πνεύμα και στην ε, συνεργασία του κυρίου Αρλάκη. Έγιναν πολλές ε, βελτιώσεις και χαίρομαι που αναφέρονται και τα δικαιώματα των γυναικών και της ε, κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά το κράτος δικαίου και η ανάγκη οικοδόμησης θεσμών, οι διάφορες προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ και υποστηρίζω τις τροπολογίες του κυρίου Κασουλίδη και τις προστίκες που προτείνει ο κύριος Κασουλίδης για την τροπολογία 173, όπου μιλάει για την ανάγκη αύξησης ε, συμμετοχής ε, των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων της ε, αρχών των Αυγανών. Αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος φυσικά της, ε, του κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό αυτό. Επισκέφθηκα το Αφγανιστάν το 2008 και το διαπίστωσα και συμφωνώ επίσης με τη συμβιβαστική παρεθμό 10. Και πάλι του κυρίου Κασούλη αναφορικά με τις ε, λανθασμένες, ε, λανθασμένους υπολογισμούς που είχαν γίνει στην αρχή. Ευχαριστώ τον κύριο Κασουλίδη που προτείνει την τροπολογία αυτή και χαίρομαι που κάποιος τόσο έξυπνος και ικανός ε, ασχολείται με το θέμα αυτό. Πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι ήταν το 2008 που ασχοληθήκαμε με το Αφγανιστάν να πω ότι αυτό που δεν μου αρέσει είναι το εξή. Η συμβιβαστική 16, αυτή η αναφορά για να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ε, ηγετικό ρόλο του στο θέμα. Δεν νομίζω ότι αυτό επιθυμούν οι Αφγανοί. Δεν νομίζω ότι το αξίζει, αυτό αξίζει στην, ε, στο Αφγανιστάν. δεν ασκούμε ε, κριτική, ε, δεν είμαστε επικριτικοί στη στάση μας, ακολουθούμε απλά τους Αμερικανούς. Και αυτή ήταν η στρατηγική μας σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να δείξουμε λίγο περισσότερη μετριοφροσύνη και να μην αναφέρουμε τόσο ξεκάθαρα ότι θέλουμε να έχουμε ηγετικό ρόλο Αν μπορούμε να συνεισφέρουμε, να το κάνουμε. Αλλά προφανώς δεν είμαστε ηγετικοί στο ρόλο μας. Είναι σημαντικό επίσης, σύμφωνο, ίσως στην συμβαστική 25, Σημαντικό λοιπόν είναι να υποστηρίξουμε την ε, πολιτική διαδικασία. Γιατί δεν είναι μόνο στρατιωτική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και η σχετική πολιτική εξέλιξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε και σε ό,τι αφορά τη σχέση με το Πακιστάν. Γιατί όλο και πιο έντονα βλέπουμε ότι είναι έντονη η συμμετοχή του Πακιστάν και αποτελεί, αν θέλετε, τμήμα του προβλήματος στο Αφγανιστάν να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο Αφγανιστάν όσο παραμένει η κατάσταση όσο έχει στο Πακιστάν και προφανώς ε, υπάρχουν στενές σχέσεις ε, του στρατιωτικού με του Ταλιμπάν και το Πακιστάν σε ό,τι αφορά την Ινδία. Ε, η κατάσταση μάλλον με το Πακιστάν και την Ινδία εμποδίζει περαιτέρω πρόοδο στο Αφγανιστάν. Να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους για την κατάρτιση των τροπολογιών αυτών των συμβαστικών. Κόντις. Ah, Α, Λάθος. Λάθος όνομα είχα γραμμένο. Κύριος Χατζηγεωργίου. Παρότι επαναλήφθηκε πάρα πολλέ φορέ, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ξαναλεχθεί ότι ο κύριο Αρλάτση έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Τόσο καλά θεμελιωμένη, που νομίζω ότι αυτή η ομόθυμη, σχετικά ομόθυμη υποστήριξη προέρχεται και από μια αδυναμία να συγκρουστούν κάποιοι με το περιεχόμενο της έκθεσης και γι' αυτό υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες τείνουν σε κάποιο βαθμό να αναιρέσουν ουσιαστικά στοιχεία της έκθεσης και εγώ θα παρακαλούσα εδώ τον κύριο Αρλάτσι να παραμείνει ε, πάνω στην ουσία της ε, δικής του έκθεσης ε, και να μην υιοθετήσει εισηγήσεις οι οποίες αναιρούν, παρά την, επαναλαμβάνω, ομόθυμη υποστήριξη, αναιρούν σε κάποιο βαθμό το περιεχόμενο της. θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στο ότι το Αφγανιστάν είναι κράτος και έχει δικαίωμα στην κυριαρχία του. Προβλήματα υπάρχουν και έχει εισηγήσει η έκθεση, τις οποίες πρέπει να στηρίξουμε. Όμως διαφωνώ προσωπικά με εισηγήσει που αναφέρουν για παράδειγμα ότι η εξάλληψη της φτώχειας το κόστος για την εξάλληψη της φτώχειας του Αφγανιστάν αντιστοιχεί στο κόστος πέντε ημερών πολέμου. Είναι μια φράση η οποία συγκλονίζει. Υπάρχει μια τροπολογία για αφαίρεση και θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Υπάρχει στην παράγραφο 13 αναφορά ότι το κόστος των πολεμικών επιχειρήσεων για μια εβδομάδα θα χρηματοδοτούσε 6.000 σχολεία γιατί να αφαιρεθεί αυτή η παράγραφος. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι στην παράγραφο 26 θα μπορούσαν τελικά να χρηματοδοτούν τους Ταλιμπάν μέσω των φορέων που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους. Δεν πρέπει να αναιρεθεί αυτή η παράγραφος. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες. Έχει και αρνητικά έκθεση και εμείς καταθέσαμε τροπολογίες οι οποίες θα τεθούν στην βάσανο και του κυρίου Αρλάτσι και της ε, Επιτροπής Εξωτερικών και της Ολομέλειας. Κλείνω λέγοντας ότι όσοι επί της ουσίας έχουν διαφωνίες για την έκθεση ε, ας έχουν το θάρρος να το πούν δημόσια παρά να επιχειρούν μέσα από ε, μια ε, τυπική υποστήριξη αλλά με τροπολογίες που την αναιρούν να, να την αναιρέσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σε χαρώ τον Πίνο Αρλάκη για την γενναία του απόπειρα. Είναι παράδειγμα ενός καλού ανθρώπου που προσπαθεί να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο σε μια δύσκολη περιοχή του κόσμου προτείνοντας ε, πολιτικές για να διορθωθούν τα λάθη ενός μακροχρόνιου πολέμου που δεν έχει φέρει και πολλές επιτυχίες παρόλο που ο Αμερικανός στρατηγός ε, μίλησε για τα πράγματα που παίρνουν θετική τροπή. Εγώ έχω αρκετές επιφυλάξεις όπως, ως προς τις πολιτικές υποδομές της χώρας που είναι πολύ επιστοδρομικές ε, και θα πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες για, για αυτήν την ανοικοδόμηση των πολιτικών υποδομών μιας χώρας που ποτέ δεν ήταν ουσιαστικά μέλος της ε, ε, παγκόσμια κοινότητα των προηγμένων χωρών. Είναι οπισθοδρομική αυτή η χώρα, γεωργική, αρκετά καθυστερημένη. Καλύτερη εποχή ήταν όταν ε, είχε βασιλέα. <laughs> Καλύτερη εποχή μιας καλοήθους μοναρχίας κατά κάποιο τρόπο, αλλά εδώ και δεκαετίες έχει φύγει ο βασιλιάς. Συμφωνώ με πολλές από τις στάσεις του εισηγητού. Έχω κάποιο πρόβλημα με κανένα δυο συμβιβαστικές τροπολογίες, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες 14, 15, 16 και κατά πάσα πιθανότητα και τις συμβαστικές 22 και 25. Βέβαια έχει κάποια ίχνη αλήθειες, αλλά Δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο αυτό των τροπολογιών και συμφωνώ με την Άννα Γκόμες ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι πολύ σημαντικά αλλά δεν αρκεί αυτό νομίζω η αναγνώριση αυτού του γεγονότος για την ανασυγκρότηση της αυγανικής κοινωνίας. Πραγματικά είναι ένα τιτάνιο έργο για οποιονδήποτε να προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει ένα έθνος που εδώ και χρόνια κατακαιρματίστηκε και καταβαραθρώθηκε από δεκαετίες βίας, λαθρεμπορή ναρκωτικών, διαφθοράς. Η διαφθορά έχει φτάσει στα υψηλά κλιμάκια τη κυβέρνηση, αυτό είναι αναφυσβήτητο και ε, ένα μεγάλο τμήμα των ε, κονδυλίων των φορολογουμένων μας ε, καταλήγει δυστυχώς σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και γίνεται αντικείμενο υπεξαίρεσης και κακής χρήσης. βέβαια, αν αποσυρθούν οι συμμαχικέ δυνάμεις, ε, υπάρχει κίνδυνος να αναλάβουν αυτό το αποσταθεροποιημένο Αφγανιστάν ή Ταλιμπάν. Οπότε θα υπάρχει και κίνδυνος και πυρηνική ε, σύρεξη μεταξύ ε, Αφγανιστάν και Ινδίας, ταλιμπανοποιημένο Αφγανιστάν και Ινδίας, που θα έχουν και πυρηνικά όπλα. Νομίζω ότι γι' αυτό αξίζει να παραμείνουμε εκεί. Παρ' όλα αυτά, ε, συμφωνώ με τις γενικές γραμμές της έκθεσης, αν και θα καταψηφίσουμε ορισμένε συμβαστικές τροπολογίες. Ωραία, δεν έχω κάποιον άλλον ε, στο κατάλογο των ομιλωτών, επομένως να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για να κάνει τα τελικά του σχόλια και μετά θα δούμε το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ κύριε Αρλάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ήταν δύσκολο ήταν δύσκολο όχι μόνο να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει, αλλά να βρούμε και ένα κοινό έδαφο στο Κοινοβούλιο, κάποιο κοινό παρανομαστή για ορισμένα στοιχεία τη έκθεση. Σε τελική ανάλυση όμω και μετά από όλε τι συζητήσει και την επεξεργασία των τροπολογιών, καθώ και την εκπόνηση των συμβιβαστικών τροπολογιών, δεν θα έλεγα ότι είναι μια έκθεση ελαχίστων και μια έκθεση που περιορίζεται απλώς σε κοινό παρανομαστή, σε ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Γιατί όλοι φυσικά προσπαθήσαμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όλες οι πολιτικές ομάδες έκαναν προσπάθεια να συμφωνήσουν για τα βασικά στοιχεία της έκθεσης και νομίζω ότι οι αδρές γραμμές ε, και η γενική της κατεύθυνση διαφυλάχθηκαν. Δεν ήταν καθόλου εύκολο και υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες σε αυτή τη συμφωνία. Πάντως νομίζω ότι η έκθεση γενικώ είναι ισορροπημένη και δεν ε, αμφισβήτησε κανείς αυτό το χαρακτηριστικό. Το ΕΛΚ ζήτησε ε, να λάβουμε υπόψη τη σημασία που έχει η στρατηγική της χώρας κατά της ανταρσίας. Δεν έχω αντίρρηση, γιατί αυτή η στρατηγική καταπολέμησης της ανταρσίας στηρίχθηκε σε μία ανάλυση που συμπίπτει και με τη δική μου. Την ανάλυση της έκθεσης. Είπα ότι όταν το περασμένο Φεβρουάριο πήγα στο Αφγανιστάν, πραγματικά έμεινα ευρόντιτος, γιατί και η ΑΕΣΑΦ ε, συμμεριζόταν την ε, ανάλυση μου και εστερνίζονταν τις επικρίσεις μου. Και είπε και η Σάφα ότι όντως χάσαμε την υποστήριξη του κοινού γιατί δυστυχώς υπήρχαν πολλά θύματα από τον άμαχο πληθυσμό. Σκοτώσαμε πολλούς άμαχους. Η στρατηγική μας λοιπόν ήταν εσφαλμένη, το παραδεχόμαστε, άρα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά, να μεταμορφώσουμε τη στρατηγική. Και το άγχος μας δεν είναι απλώς να μειώσουμε τα θύματα του άμαχου πληθυσμού, είναι να μην έχουμε καθόλου θύματα άμαχου πληθυσμού, να έχουμε μηδέν απώλειες και να ξανακερδίσουμε την ε, εμπιστοσύνη του κοινού με μια στρατηγική που θα είναι συνδυασμό πολιτικής και στρατιωτικής επέμβασης. Οπότε αυτή η ανάλυση για την κατάσταση του Αφγανιστάν τη συμμερίζονται και οι συμμαχικές δυνάμεις του Αφγανιστάν. Αυτό ό,τι αφορά το επικριτικός ή το κριτικό τμήμα της έκθεσης, αλλά νομίζω ότι είναι και επικοδομητική έκθεση, γιατί αναφέρεται και στα θετικά στοιχεία και που θα πρέπει να επικεντρώσουμε στο μέλλον τη στρατηγική για το Αφγανιστάν. Δεν θα προσπαθήσουμε εμείς να συγκροτήσουμε όλες τις πτυχές του Αφγανιστάν. Αν αρχίσουμε να ε, φιλοδοξούμε ή να αξιώνουμε ότι θα πρέπει το Αφγανιστάν να αναβαθμιστεί σε όλες τις λεπτομέρειες και τις πολιτικές οικονομικές. Δεν θα το αποφασίσουμε αυτό εμείς. Η αφγανική κοινωνία θα το αποφασίσει. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε τρία-τέσσερα σημεία. Και για τα σημεία αυτά θα... Στα σημεία αυτά θα συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες και τα δαψιλή κονδύλια που στέλνουμε προς το Αφγανιστάν. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να εμείνω σε τέσσερις άξονες στην έκθεση. Έγινε μια πολύ σημαντική προσθήκη από τον κύριο Νόιζερ και τη σοσιαλιστική ομάδα για το θέμα το... της δικαστικής εξουσίας, του δικαστικού κλάδου. Ήταν όντως μια παράληψη της έκθεσης. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μια σοβαρή εκπαίδευση αστυνομική δύναμης αν δεν έχουμε παράλληλα μια λειτουργούσα δικαστική εξουσία που θα ε, εγγυάται το σεβασμό του κράτους δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ και το δικαστικό κλάδο. αλλά δεν πιστεύω θα πρέπει να επεκταθούμε στη γενική ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν. Και εκεί έγινε η βασική διαφορά με το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η έκθεση εκείνη είναι πολύ πιο πολιτική, επισέρχεται σε πολιτικά θέματα, με την, έκθεση με την ελευθερία που χαρακτηρίζει τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Δεν υπησέρχεται σε πολιτικά θέματα, δεν επισέρχεται σε βασικά στοιχεία. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο βρίσκεται εδώ για να είναι πιο ευρύ και γενικώ τη του και πιο ελεύθερο. Σε ό,τι αφορά τι παρατηρήσει του κυρίου Κασουλίδη για την ε, κατάργηση, ε, εξάλληψη της καλλιέργειας ε, των οποίων φυτών στο Αφγανιστάν. Έχω μια τροπολογία που προτείνω στην αφγανική κυβέρνηση να απαγορεύσει δια νόμου τη χρήση χημικών παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων στο Αφγανιστάν. Αυτό έκανε και ο ΙΕ στη Βολιβία και το Περού. Έτσι μπόρεσαν αυτές οι δύο χώρες να μειώσουν τις, την καλλιέργεια το, της κόκας και Κάτι που δεν ισχύει στην Κολομβία που χρησιμοποιούνται χημικά φυτοφάρμακα για την εξουδετερώση των καλλιεργειών. Ο κύριος Κασουλίδης είναι κατά της χρήσης φυτικών φυτοφαρμάκων και εγώ συμφωνώ. Θα πρέπει να γίνεται με το χέρι η εκρίζωση των οποίουχων φυτών στο Αφγανιστάν. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χημικά μέσα, χημικά φυτοφάρμακα για κάτι τέτοιο. Τα χημικά φυτοφάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί στο Αφγανιστάν, αλλά παρόλα αυτά ήταν αποτελεσματικά. Είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν είχαν αποτέλεσμα, δεν, χρησιμοποιη... δεν είχαν επιτυχία. Δεν υπάρχει όμως εγγύηση ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτά που έγιναν πριν από μία τριακονταετία, που ούτως ή άλλως κατηγορήθηκαν από τον ΟΗΕ, γιατί είναι ένας τρόπο για να αυξηθεί ε, η εχθρότητα, η τρομοκρατία. Χρειάζεται μια πενταετία για να εξαλειφθεί η καλλιέργεια των φυτών, χρησιμοποιώντας και, και ένα μικρό τμήμα των, της ε, ευρωπαϊκής Χωριές και δωρεών προς το Αφγανιστάν. Και αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Η έκθεση προτείνει τη σύσταση και ενός ειδικού σώματος για την ανάληψη αυτού του καθήκαντος, γιατί ο Αφγανός υπουργό καταπολέμησης των ναρκωτικών δεν είναι αρμόδιος ούτε κατάλληλος για να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα ειδικό σώμα που θα παρτίζεται και από Αφγανούς αλλά και από τεχνική υποστήριξη της παγκόσμιας κοινότητας και κάλλιστα μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε μία πενταετία. Μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει ουδέποτε στο Αφγανιστάν. Και αυτή είναι και η βασική, από τι βασικέ επικρίσει τη έκθεση. Δέκα χρόνια μετά, κανεί δεν κατήρτισε ένα συνολικό και σοβαρό σχέδιο για την εξάλληψη της ε, καλλιέργειας της Μύκονος της Υπνοφόρου, τη οποίου παπαρούνα. Και χαίρομαι που οι πολιτικές ομάδες τελικά συμφωνούν με την ανάλυση αυτή και δεν ε, κατέθεσαν τροπολογίε για το σημείο αυτό. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για το Αφγανιστάν όταν θα εγκριθεί αυτή η έκθεση. Τέλος, για τα σχόλια του ΕΛΚ. Ήταν πολύ επικοδομητική στάση του σκιώδου συγητού και θα ήθελα και εγώ να ε, συγχαρώ τον κύριο Κασουλίδη και τους υπόλοιπους σκιώδους συγητές για τη συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας καθ' όλη τη διάρκεια τη διαπραγματευτική διαδικασία. Συντρέχουν οι προποθέσει λοιπόν να συγκεντρώσουμε ευρεία συνένεση για την έκθεση. Φυσικά υπάρχουν και τροπολογίε που προσπαθούν να παλύψουν σημαντικά τμήματα. Το θέμα τη ε, κατάσταση των γυναικών, εκλογές, ε, συνέπειες της παγκόσμιας ενίσχυσης. Εγώ εξέφρασα τη γνώμη μου, αλλά άφησα ψηφοφορία κατά το δοκού. Να ψηφίσουμε να δούμε ποια θα είναι η κρατούσα γνώμη. Κύριε Τάλερ, σας ευχαριστώ που είπατε ότι το μήνυμά μας θα πρέπει να είναι σαφές. Γιατί πραγματικά έτσι θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με σαφήνεια και θα φροντίσουμε να εφαρμόσουμε σωστά τις συστάσεις της έκθεσης και είναι σημαντικό από τώρα να μεριμνήσουμε ώστε όλο το έργο που επιτελέσαμε τον προηγούμενο χρόνο να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πολιτική λύση. Φυσικά αυτό λέει και η έκθεση. Είναι συνέχεια της ε, διαδικασίας της Καμπούλ και της διάσκεψης του Λονδίνου εκεί αναφέρθηκε με σαφήνεια ότι δεν είναι δόκιμη στρατιωτική λύση στο Αφγανιστάν. Και αυτή είναι και η συνέχεια της διαδικασίας Καμπούλ. Είπατε ότι η τροπολογία 273 δεν έλειφθη δόντως υπόψη. Η τελευταία όμως συμβεστική λύση, η υπαριθμόν 25-26 που δέχτηκε και ο κύριος Νόιζερ μιλούν για ανάγκη σταδιακής αποχώρησης των συμμαχικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Έχουμε και την έκθεση Μπάγκλ που προβλέπει διορία διετή για την αποχώρηση όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα ψηφίσουμε για αυτές. Πάντως, δεν νομίζω ότι οι συμβαστικές λύσεις συνιστούν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Δεν συμβιβαστήκαμε Απλώς προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ισορροπία και τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Κυρία Γκόμες, δεν σας άρεσε αυτό που λέμε για τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον ηγετικό ρόλο που αξίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι συμβαστικές τροπολογίες αναφέρονται στην UPOL. Οι τροπολογίες για την δεν αναφέρονται στο ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει το ηγετικό ρόλο που της αξίζει στο θέμα της εκπαίδευσης της αστυνομίας, των αστυνομικών δυνάμεων. Συμφωνώ ότι <laughs> σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ηγήθηκε της διαδικασίας, δεν ηγήθηκε της διαδικασίας. Γι' αυτό δεν θέλουμε νέα στρατηγική. Δεν θα ξοδεύαμε τόση ενέργεια να καταρτήσουμε τη νέα στρατηγική. Εγώ θα ήμουν τελευταίο που θα έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ηγετικό ρόλο μέχρι τώρα στο Αφγανιστάν. Οπότε αυτό που λέμε για τον ηγετικό ρόλο θα ήθελα να το ερμηνεύσετε συσταλτικά σε αυτό που ζήτησε η κυρία Γετενμάκη δηλαδή για τη Γιούπολ. Σε ό,τι αφορά το Πακιστάν δίκιο έχετε ότι έχει κέριο ρόλο να διαδραματίσει η χώρα αυτή. Αλλά αν ακούσετε τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, θα διαπιστώσετε ότι είπε πολύ σημαντικά πράγματα που ευθυγραμμίζονται πλήρω με αυτά που είπατε εσεί. Φυσικά χρειαζόμαστε και τη συνεργασία του Πακιστάν και έχει δικαίωμα το Πακιστάν να εκφέρει γνώμη για το Αφγανιστάν. Μην ξεχνάτε ότι το Πακιστάν έχει σύνορα 3.000 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν. Το ίδιο και το Ιράν. Έχει εκτενέστατα σύνορα με το Αφγανιστάν. Οπότε αυτές οι δύο χώρες, Ιράν και Πακιστάν, έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη για το Αφγανιστάν και είναι οι πρώτες χώρες που θα πρέπει να δώσουν τη γνώμη τους. Γιατί μιλάμε για την ε, πακιστανική την ιρανική επέμβαση στο Αφγανιστάν. Κατά τη γνώμη μου είναι ε, αδόκιμη αδόκιμος αυτός ο χαρακτηρισμός. Φυσικά, μια χώρα που έχει σύνορα με μια άλλη χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, έχει δικαίωμα να εκφέρει γνώμη και να υποβάλει και πρόταση. Υπάρχουν και μερικές τροπολογίες για την περιφερειακή λύση με ανάμειξη του Πακιστάν, του Ιράν, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό τμήμα Βέβαια δεν στήριξα την έκθεσή μου σε αυτό το θεμέλιο γιατί το ζήτημα είναι εξαιρετικά πολύ σύνθετο και περίπλοκο και θα μας παρασύρει σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια έκκληση. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρχαν κάποια ψήγματα αυτή της στρατηγικής, αλλά δεν είχε αναλυθεί καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Χατζηγεωργίου, Σας ευχαριστώ για την εκτίμησή σας προς την έκθεση. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Νομίζω ότι ήταν πολύ έντιμες οι συμβαστικές τροπολογίες και σεβάστηκαν τα βασικά στοιχεία της έκθεσης και αυτή είναι η διαδικασία η κοινοβουλευτική. Και όντω τα πράγματα είναι δύσκολα μερικέ φορέ, αλλά αυτό είναι το έργο μα. Το κόστο του πολέμου που λέτε, όντω έχετε δίκιο. Αλλά αυτό που με προβλημάτισε και θα να σα ρωτήσω, γιατί όλε σχεδόν οι ομάδε ήταν κατά των δύο παραγράφων εκεί που μιλάω για το κόστο για το κόστος του πολέμου που λέμε ότι το κόστος του πολέμου στο Αφγανιστάν θα ε, ε, ήταν τόσο μεγάλο που θα μπορούσαμε το, να το χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο και να ξεριζώσουμε τη φτώχεια στον κόσμο. Περισσότερες α, ε, ομάδες ήταν κατά της φράσης αυτής και ήταν τόσο συντριπτική πλειοψηφία κατά των παραγράφων αυτών που χρειάστηκε να τις α, ε, αποσύρω. Αλλά πραγματικά γιατί όλοι έπεσαν να με φάνε με αυτόν τον υπολογισμό. Υπάρχουν και άλλες παράγραφοι στην έκθεση που αναφέρονται ρητά στο τεράστιο κόστος, δυσβάσταχτο κόστος του Αφγανικού πολέμου. Είναι λογικό να συγκρίνουμε το κόστος αυτού του πολέμου με εναλλακτικέ λύσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε εφαρμόσει πριν από μία δεκαετία, για παράδειγμα. Εναλλακτικέ λύσεις, όχι στρατιωτικές και πολεμικές. Και να δούμε όλα αυτά τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για τον πόλεμο, πώς θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί όλου. Εν πάση περιπτώσει, μια ναι, και υπήρξε σχεδόν ομοφωνία εις βάρος αυτών των παραγράφων, αναγκάστηκα να τις ε, περικόψω κι εγώ. Και παρόλο που εγώ επί της ουσίας είμαι αντίθετος και ήμουν υπέρ αυτού του υπολογισμού. Κύριε Τάνοκ, σας ευχαριστώ για, για τα καλά σας λόγια. Όντως δεν ήταν καθόλου εύκολο να συγκεράσω όλες αυτές τις διστάμενες απόψεις. Αλλά μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί είστε κατά ε, των τροπολογιών που αναφέρατε. Μπορούμε και κατηδίαν ε, να, το εξετάσουμε για να το καταλάβω κι εγώ. Δεν ήσασταν στι διαπραγματεύσει όταν συντάξαμε τι συμβαστικέ τροπολογίε και λυπούμε γι' αυτό, γιατί τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να τι συζητήσουμε και να δούμε που είχατε αντιρρήσει για να εξασφαλίσουμε και τη δική σα υποστήριξη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για την παρέμβασή τους. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 9 Νοεμβρίου και το Δεκέμβριο το θέμα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Πέρα στη συνεδρίασης, ένα-δυο λεπτάκια διάλειμμα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρίου για να μπορέσουν να αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν πλέον δουλειά στην αίθουσα. Ευχαριστώ.